Οι αρμόδιε βελγικέ αρχέ με ενημέρωσαν ε, για την εκλογή του κυρίου Μάρκ Ντέμεσμάκερ από 1η Φεβρουαρίου του 2013. Να ρωτήσω κατά πόσο αυτό ισχύει. Μισό λεπτό. Όχι. Οι αρμόδιες βέλγικες αρχές με ενημόρισαν για την εκλογή του κυρίου Μάρκ Ντέμεσμάκερ από 1η Φεβρουαρίου 2013 αντικαθιστά την κυρία Φρίντα Μπερέπουλς. Ε, σας καλωσορίζω και να σας υπονθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου υπό τον όρο ότι θα υπογράψει ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα το οποίο δεν συνάδει με το αξίωμα του Ευρωβουλευτή. Οι αρμόδιες ε, πολωνικές αρχές με ζήτησαν να άρω την ε, ασυλία του κυρίου Τζάτσεκ Κούρσκ σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγραφός 2 του κανονισμού το αίτημα αυτό ε, απεστάλησε στην Αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας ενημερώσω ότι